Okay, dear colleagues, ladies... Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, είναι 3 και 5 και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Είναι τα, από όσο ξέρω, είναι η τελευταία μας συνεδρίαση της Επιτροπής μας σε αυτή την νομοθετική θητεία, οπότε μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρκετά επιτυχής μάλιστα Πετύχαμε πολλά όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και όσον αφορά πολύ σημαντικά ε, εμπορικά νομοθετήματα. Η Επιτροπή Ίντα λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί ότι κλείνει τις εργασίες της με περηφάνεια. Κοιτώντα πίσω στην τελευταία πενταετία παρόλα αυτά, σε αυτή την τελευταία συνεδρίαση δεν θα τεμπελιάσουμε. Ε, υπάρχει λοιπόν και το σχέδιο ημερήσιας διάταξης προτείνω να προσθέσουμε μετά το σημείο 6 ένα νέο σημείο τι τελευταίε εξελίξεις στον ΠΟΕ για την διευθέτηση διαφορών. Υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να αλλάξει κάτι στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Ωραία, λοιπόν με αυτή την προσθήκη υιοθετούμε την ημερήσια διάταξη. Πάμε στο σημείο 2, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων, τη συνεδρίαση της 18 η Μαρτίου. Έχουμε τα πρακτικά στα χέρια μας, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα υιοθετηθούν. Σημείο 3, ανακοινώσεις του Προέδρου όπως ε, συνήθως ε, μεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση σε όλη την Ευρώπη οπότε καλωσορίζουμε και τους ε, ανθρώπους που κάθονται στις οθόνες από το Λιονεμπουργκ μέχρι τη Λισαβόνα, από το Ελσίνκι μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από τη Βαρσοβία μέχρι το Παρίσι. Καλώς Για να διευκολυνθεί η διερμηνία παρακαλούμε να μιλάτε με κανονική ταχύτητα, καθαρά και δυνατά. Δεύτερο σημείο της ημερήσιας ε, διάταξης, ε, οι πληροφορίες ε, της, των εισηγητών για την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Ο κ. Σάντι και εγώ στείλαμε μια επιστολή στην Ρουμανική Προεδρία ζητώντας πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα αυτής της συμφωνίας και προς το παρόν δεν έχουμε λάβει απάντηση. Αλλά ακούμε φήμες ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής πρόκειται να λάβει χώρα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα, όπου σημαίνει ότι θα ασχοληθεί με αυτή τη συμφωνία το νέο κοινοβούλιο πλέον. Και θα ανακοινωθεί στην πρώτη συνεδρίαση πιθανότητα του νέου κοινοβουλίου. Τρίτον, έχω μια θλιβερή είδηση. Ένα από τα πιο έμπειρα μέλη της γραμματείας δυστυχώς ε, μας εγκαταλείπει. Ήταν το δεξί χέρι του Αλμπέρτου και του Μάρτιν. Ήταν μια ζωντανή εγγύηση που είχα εγώ ως πρόεδρος την τελευταία πενταετία ε, διασφάλιζε την καταπληκτική προετοιμασία των συνεδριάσεων που με καθησύχαζε εμένα, δεν είχα κανένα άγχος, κανένα πρόβλημα. Πάντα ομαλά πρόεδρευα τη συνεδρίας εδώ της Επιτροπής ε, χάρη σε αυτήν, οπότε ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας, ε, για τα πολλά χρόνια που μας βοηθήσατε εδώ στην Επιτροπή και σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον. δεν μπορώ να φανταστώ καν πώς θα οργανώνουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας χωρίς εσάς, αλλά κάπως θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ και σα εύχομαι ότι καλύτερο. Point Σημείο 4. Σύναψη της Διεθνούς Συμφωνίας ε, για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζες ελιές του 2015. Η εισηγήτρια είναι η Ελεονόρα Φορέντσα και θα της δώσω αμέσως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Διεθνή Συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζες ελιές του 2015 ακολουθεί την Συμφωνία του 2005 τον Νοέμβριο του 2013. Το Συμβούλιο έδωσε έγκριση στην Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ένωσης εν ώψη μια νέα διεθνού συμφωνία για το ελαιόλαδο και τι επιτρέπεζε ελιέ. Κατά τη διάσκεψη στη Γενέβη των Ηνωμένων Εθνών ε, τον Οκτώβριο του 2015, εκπρόσωποι των 24 κρατών μελών τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη και δύο ε, διακυβερνητικοί οργανισμοί συνέταξαν το κείμενο της Νέας Συμφωνίας. Η Διεθνή Συμφωνία για το Ελαιόλαδο και τις Επιτραπεζές Ελιές υπογράφηκε εξ ονόματος της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης της 28 Νοεμβρίου του 2015 στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με επιφύλαξη συνάψη και ολοκλήρωση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η νέα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Μεταξύ των στόχων της συμφωνίας αυτής ε, έχουμε την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας γεωργίας, ευνόηση του συντονισμού των πολιτικών παραγωγής, βιομηχανοποίηση, αποθήκευση και διάθεση στο εμπόριο του ελαιολάδου, του πυρενελαίου και των επιτραπέζων ελιών. Ενθάρρυνση της έρευνας και της ανάπτυξης και ευνόηση των, σε μεταφοράς τεχνολογίας και δραστηριοτήτων εκπαίδευση στον τομέα της ελαιοπαραγωγής. Η συμφωνία ε, θεσπίζει ένα όργανο αποφάσεων, συμβούλιο των μέλων όπως ονομάζεται, που θα ασκεί όλες τις εξουσίες ε, και όλες τις απαραίτητε λειτουργίες για την εφαρμογή των στόχων της ε, συμφωνίας. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το Συμβουλίο των Μελών μπορεί να τροποποιήσει τις εκχωρήσει και τις ονοματολογίες ε, των ελαιών, των επιτραπέζιων ελαιών και των πυρηνέλαιων και συνεπώ να τροποποιήσει την συμφωνία δεδομένου ότι η ελαιοπαραγωγή αποτελεί ένα σημαντικό τομέα για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία και της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και της Ιταλίας, ε, αποτελεί ένα προϊόν ε, υψηλότερη σημασία για την Ευρώπη και έτσι ζητάμε ευνοϊκή αντιμετώπιση από το Κοινοβούλιο όσον αφορά αυτή τη συμφωνία, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να συμβάλλει δραστήρια στην διεθνή συνεργασία για το ελαιόλαδο και τι τη ελιάς. Ωστόσο, θλίβομαι για τις καθυστερήσεις της μεταφορές παρούσας ε, συμφωνίας ε, στο Κοινοβούλιο και την έλλειψη έγκαιρων πληροφοριών από άλλα θεσμικά όργανα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είναι πολύ σημαντικός ε, ο τομέας αυτός της ελαιοπαραγωγής, ειδικότερα για την Ευρώπη της Μεσογείου και για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει την κρίση. Σκεφτείτε τι γίνεται στην Νότια Ιταλία αυτή τη στιγμή στην Απούλια μετά από την παγωνιά και την ξύρανση κάποιων ελαιόδενδρων. Έχουμε μια δραματική κρίση στην ελαιοπαραγωγή που είναι χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής. Ε, οι διεθνεί συμφωνίε που σχετίζονται με την κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται στην συνένεση του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το λόγο, Καλό το Συμβούλιο και την Κομισιόν να ενημερώνουν επαρκώ ε, το Κοινοβούλιο, ειδικότερα όσον αφορά οποιαδήποτε απόφαση που θα μπορούσε να ληφθεί σε σχέση με το άρθρο 4 τη απόφαση του Συμβουλίου. Ε, οι διεθνείς συμφωνίες υπόκειται στη δεσμευτική ψηφοφορία του Κοινοβουλίου, η εφαρμογή τους ακόμα και αν είναι προσωρινή δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συνένεση του Κοινοβουλίου στο μέλλον. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να λαμβάνει έγκαιρα λεπτομερείς πληροφορίες αντίστοιχες με εκείνες που παρέχονται στο Συμβούλιο, ειδικότερα όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συμβουλίου των μελών όπου θεσπίζει η Συμφωνία. Πέραν αυτού, όταν το Συμβούλιο των Μελών καλείται να υιοθετεί τροποποιήσεις στις ονοματολογίες ε, των διαφόρων προϊόντων ε, σύμφωνα με τα παραρτήματα Β και Γ ε, τη συμφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 19, η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την θέση που θα λαμβάνει εξ ονομάτων τη Ένωση. Πρόσφατα ξεκίνησε μια συζήτηση μετά από πρόταση των Ιταλικών Ενώσεων για το ενδεχόμενο αλλαγή ορισμένων παραμέτρων για το έξτρα παρθενό ελαιόλαδο ώστε να μειωθεί το όριο οξύτητας από το 0,8% στο 0,5% και θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Η Επιτροπή Άγκρη στην ογνωμοδότησή τη πρότεισε μια υπόθεση εργασία για την εισαγωγή μια νέα ονομασία, μια νέα κατηγορία ε, του έκτρα παρθένου ελαιολάδου υψηλή ποιότητα. Μα φαίνεται ένα ενδιαφέρον σενάριο το οποίο θα βοηθήσει να προστατεύσουμε καλύτερα τι ποιοτικέ παραγωγέ. Επίση, θεωρώ την αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εργαστεί στο πλαίσιο τη συμφωνία για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ελαιοπαραγωγών χωρών, ώστε να διασφαλίζονται τα μέγιστα πρότυπα ποιότητα και η πλήρη συχνηλασιμότητα, ώστε να εφαρμόζεται επαρκώ η αρχή τη διαφάνεια ενώπιον των καταναλωτών και να αποφεύγονται οι απάτε στον τομέα. Θα θέλαμε τέλο να ζητήσουμε από την Κομισιόν να ξεκινά μια απλοποιημένη διαδικασία ε, δυνάμει του άρθρου 18 ε, παραγράφου 9 της Συνθήκης Λειτουργίας ε, για τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συμβούλιο των Εταίρων. Όπω υποβλήθηκε και στο Κοινοβούλιο για τη συνένεσή του, κατά την άποψή μα, οι θέσει που θα πρέπει να εκφράζονται εξ ονόματο τη Ένωση σε οργανισμού που θεσπίζουν διεθνεί συμφωνίε θα πρέπει να αποφασίζονται από το Συμβούλιο μετά από πρόταση τη Κομισιόν χωρί δυνατότητα απλουστευμένη διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2018, παράγραφο 10. Δεν είναι σαφές ακόμα αν αυτή η πρόταση ισχύει ακόμα ή αν έχει αποσυρθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές και στην κυρία Σάιφη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ εξ του ονόματο του συναδέλφου Φερνάντο Ροά, ο οποίο δεν μπορεί να παρευρεθεί <coughs> σήμερα και μου ζήτησε να διαβάσω την παρέμβασή του ω σκιώδη εισηγητή του ΕΛΚ. Η παρέμβασή του είναι η εξή. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα τη χαρά να συμμετάσχω στις εργασίες της Επιτροπής μας και να συζητήσουμε σήμερα την σύναψη αυτής της συμφωνίας για τις επιτραπέζιες ελιάς και το ελαιόλαδο. Είναι η πρώτη έκθεση για την οποία στην Επιτροπή ΙΝΤΑ μου ανατέθηκε να είμαι σκιώδης εισηγητής. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με λυπεί το γεγονό ότι δεν ε, επαστάλει πιο νωρί τη συμφωνία στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή, έτσι ώστε να την εγκρίνουμε πιο νωρί. Η κυρία Φορέντσα ήδη ανέφερε τους στόχους της συμφωνίας, επομένως δεν θα τους επαναλάβω. Δημιουργείται ένα όργανο λήψης αποφάσεων, αυτό το Συμβούλιο των Μελών, και είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πραγματικό χρόνο να έχει ενημέρωση για να μπορεί να γνωρίζει πώς εξελίσσεται η εφαρμογή της συμφωνίας και τι κάνει η Επιτροπή. Κλείνοντα, θα έλεγα ότι η συμφωνία αυτή είναι συμβατή με τι πολιτικέ και τι στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση και προτείνω ότι είναι. Ε, να δώσουμε την εγκρισή μας. Στη... Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους, μιας και είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε και για το έργο που επιτελέσαν όλη αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σάιφη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ομάδα ECR λοιπόν εγκρίνει ε, την ε, έκθεση της Επιτροπής και λυπάται για την ε, καθυστερισμένη λήψη των σχετικών πληροφοριών. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. τονίζοντας πως όντως βρισκόμαστε υπό μεγάλη χρονική πίεση και μετά την ε, σύσταση για ολοκλήρωση λοιπόν της συμφωνίας το 2017 όταν και υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Μόνο πριν από δύο εβδομάδες έφτασε η απάντησή τους. Γι' αυτό λοιπόν ε, πραγματικά φαίνεται πως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Η κυρία Ζήλκεμπουργκ, εκ μέρου Ευρωπαϊκή Επιτροπής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχάς πως εκτιμούμε πάρα πολύ την θετική στάση της Επιτροπής ΙΝΤΑ για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Όπως είπατε και εσείς, είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία ήδη έχει τεθεί σε ισχύ προσωρινά. Είναι λειτουργική λοιπόν, είναι όμω πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα μήνυμα στους εταίρους μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί και θα τηρήσει τι συμφωνίε της. Υπάρχουν φυσικά ορισμένε προτεραιότητες για το διεθνές εμπόριο, οι οποίες είναι αρκετά ε, σημαντικές Και είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια καλή συνεργασία η οποία θα ενισχύσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω. Η εναρμόνιση επίσης των προτύπων του IOC είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη διευκόλυνση του εμπορίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις και το χρονικό διάστημα που κράτησαν ανάμεσα σε Συμβούλιο και Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 4, το οποίο ρυθμίζει μια απλουστευμένη διαδικασία για ε, τεχνικές λεπτομέρειες και παραρτήματα της ε, συμφωνίας, είναι δυνατόν να γίνει τροποποίηση στο μέλλον. Οι συζητήσεις λοιπόν και οι διαπραγματεύσεις για αυτά τα σημεία κράτησαν πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Τώρα μόλις καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις. Και ακριβώς επειδή θέλουμε να έχουμε πλήρη διαφάνεια, όλες οι τροπολογίες, κάθε μία από αυτές, είναι στη διάθεσή σας. Όλα, όλα λοιπόν τα προσχέδια της ε, συμφωνίας, τηρώντας τους ε, κανόνες περί διαφάνειας, αποστέλλονται αμέσως στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω πως ε, είναι εγγυημένη η διαφάνεια κατά την άποψή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά να ξέρετε πως φυσικά πάντα θα ζητάμε περισσότερη διαφάνεια και καλύτερη βελτιωμένη συνεργασία ανάμεσα στα θεσμικά όργανα. Δυστυχώς όμως, διαπραγματευόμασταν επί τρία χρόνια με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την συνεργασία στις συμφωνίες που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες και το Συμβούλιο δεν ήταν σε θέση να συμβαστεί με το Κοινοβουλίο. τα ελάχιστα δικαιώματα που έχουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα έχουμε επειδή απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, κατόπιν αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό φυσικά είναι απαράδεκτο. Και ο κύριος Μπροκ και εγώ διαπραγματευτήκαμε εκ μέρου του Κοινοβουλίου και αρνηθήκαμε να ολοκληρώσουμε μια τέτοια συμφωνία με το Συμβούλιο. Αυτό βέβαια είναι καθήκον και αρμοδιότητα του επόμενου Κοινοβουλίου. Οφείλει λοιπόν να πιέσει για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που παρενέβησαν και την ε, Επιτροπή για τις εξηγήσει της. Δεν έχω παρά να επαναλάβω και εγώ ότι ανησυχούμε για την καθυστέρηση που σημειώθηκε και συμφωνώ με το αίτημα στο μέλλον να υπάρχει καλύτερη κοινοποίηση των πληροφοριών και στο Κοινοβούλιο και στη διαπραγματευτική φάση, δεδομένου ότι πρόκειται για το τελευταίο φάιλ της ΣΥΝΤΑ που θα ψηφίσουμε σε αυτή τη θητεία. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι τις ευχαριστίες μου προς όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής για την εργασία στο πλαίσιο της οποίας συνεργαστήκαμε τα τελευταία χρόνια. Thanks Ευχαριστούμε πολύ. Because Ακριβώς λοιπόν λόγω της πίεσης χρόνου πρέπει να ψηφίσουμε αύριο το πρωί στις 10. Αυτό τι σημαίνει. Αν υπάρχουν τροπολογίες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξουν, αλλά αν υπάρχουν, να ξέρετε πως προθεσμία είναι σήμερα στις 6 το απόγευμα. Και φυσικά δεν θα υπάρχει δυνατότητα μετάφρασης των τροπολογιών, εφόσον υπάρξουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ να τις υποβάλλετε όχι στα στονικά α πούμε, αλλά στα αγγλικά. Έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τις διαβάσουμε. Προθεσμία λοιπόν για την κατάθεση τροπολογιών 6 το απόγευμα σήμερα και στα αγγλικά παρακαλώ. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημείου 4 της ημερήσιας διάταξης. Και περνάμε στο σημείο 5. Να καλωσορίσω τον καθηγητή Μπάρτ Κέρμαντς. Καλώς ήρθατε ξανά. Είναι καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Λουβά. Και επικεφαλής της συντακτικής ομάδας ε, για τη μελέτη σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των εμπορικών πολιτικών στον δυτικό κόσμο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, διότι αν θυμάστε έχουμε συζητήσει διεξοδικά τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και στην ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών, αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP, αλλά και αργότερα για τη συμφωνία ΣΕΤΑ και την διάκριση των εξουσιών, την αποκλειστική και μεικτή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Συζητήσαμε επίσης και το ρόλο που οφείλουν να διαδραματίσουν οι ε, ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι λοιπόν πολλά ερωτήματα, πολύ σημαντικά. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω τον ε, καθηγητή Κέρμαντς και χαίρομαι πάρα πολύ που θα μας δώσει απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και το PowerPoint, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε να συνοψίσω τα στοιχεία και τα ευρήματα της μελέτης μας. Φυσικά δεν έκανα μόνος μου τη μελέτη. Ήμασταν μία ομάδα τεσσάρων συνεργατών ένας από αυτούς είναι ο Γιώνα Τριάσον, συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, κάθεται δίπλα μου. Και στη μελέτη συγκρίναμε τέσσερα κοινοβούλια σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους και την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν στις διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες για αυτόνομα εμπορικά μέτρα και στη μελέτη μας, εκτός από το ότι εστιάσαμε σε αυτά τα κοινοβούλια, προσπαθήσαμε να δούμε πώς ο νομοθέτης ε, δράσε υπό εθνικό επίπεδο. Στην παρουσίασή μου θα εστιάσω όχι στα αυτόνομα εμπορικά μέτρα, ούτε στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά στις υποεθνικές αρχές, στο υποεθνικό επίπεδο και ελπίζω να μου κάνετε σχετικές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τις διαφορές μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και υπάρχουν δύο-τρεις φράσεις που συνοψίζουν νομίζω την ουσία της μελέτης μας. Αυτές τις φράσεις δεν θα τις βρείτε στην ίδια την ε, μελέτη, διότι τις φύλαξα για να τις παρουσιάσω προφορικά. Αλλά ας πούμε ότι αν ήμουν βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας ή του Καναδά, θα ζήλευα. Αν ήμουν όμως μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου, θα μου ξυπνούσε την περιέργεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν ήμουν ευρωβουλευτή που ούτε ήμουν ούτε και θα είμαι υποψήφιος, αλλά φανταστείτε, αν ήμουν ευρωβουλευτή, θα χαιρόμουν μεν, αλλά θα πρόσεχα πάρα πολύ τι γίνεται δε. Συγκριτικά λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί μεγάλη επιρροή στις διεθνείς εμπορικές διαπραγματεύσεις. Στη σύγκριση λοιπόν που κάναμε μεταξύ των τεσσάρων θεσμών, το Κογκρέσο δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κοινοβούλιο του Καναδά, τη Αυστραλία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό παίκτη, ακριβώ όπω το Αμερικανικό Κογκρέσο. Αν δείτε τα τρία στάδια τη ε, διαπραγματευτική διαδικασία, το πρώτο, το στάδιο τη εντολή, είναι εκείνο όπου αποφασίζεται το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης και τα όρια που μπορούν να φτάσουν ή να μην ξεπεράσουν. Μετά έχουμε το στάδιο της διαπραγμάτευσης και το τελευταίο στάδιο είναι εκείνο της ε, επικύρωσης. Όμως το σημαντικότερο στάδιο όλης της διαδικασίας είναι το τελευταίο, το στάδιο της κύρωσης της συμφωνίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι τα βέλη δείχνουν προς τα αριστερά. Πάνε προς τα πίσω λοιπόν, διότι στη τελική ανάλυση το σημαντικό είναι αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικός παίκτη διότι δίνει την έγκρισή του. Παρομοίως, το Αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να συμφωνήσει στο αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι το σημαντικότερο από τα τρία αυτά στάδια. Εδώ υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στο Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μεταξύ αυτών των δύο και των κοινοβουλίων του Καναδά και της Αυστραλίας. Στη διαφάνεια εδώ και στις επόμενες δύο βλέπετε κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτον, βλέπετε τις θεσμικές διαφορές των τεσσάρων κοινοβουλίων. Βέβαια, η ιδιαιτερότητα των ΗΠΑ είναι ότι έχει και τη γερουσία και τη βουλή των αντιπροσώπων. Παρομοίω και ο Καναδά. Από την άλλη, βλέπετε το βέλο που είναι αμφίδραμο. Πηγαίνει και προ τα πάνω και προ τα κάτω. Προ τα πάνω, λοιπόν, όσο πιο πάνω, τόσο πιο ισχυρό το κοινοβούλιο. Όσο πιο κάτω, τόσο λιγότερο ισχυρό. Και με τα κίτρινα πλάγια γράμματα και τα κίτρινα βέλη βλέπετε αυτό που εμείς ονομάζουμε άτυπες μορφές εργασίας ή εν μέρη τυπικές, επίσημες. εσωτερικές διεργασίες δηλαδή εντό των κοινοβουλίων. Και όταν περάσουμε στο στάδιο τη εντολή, θα δείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σύγκριση με το Κογκρέσο έχει αρκετά ισχυρότερη θέση σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της εντολής. Παρότι δεν έχει επίσημα αρμοδιότητα να καθορίσει το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων σίγουρα, ασκεί μεγάλη πίεση. Και αυτό προκύπτει από τη συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου και αναφέρομαι στην ε, Συμφωνία Πλαίσιο του 2010. Βέβαια, ο, η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλεται εν μέρη και στον ε, έλεγχο που ασκεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός εταίρος ακόμα και στο στάδιο της εντολής. Και φυσικά, αυτό το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθεί να μπαίνει στο παιχνίδι ολοένα και νωρίτερα και να αντιδρά με ψηφίσματα και με διάφορους άλλους τέτοιους τρόπους όταν ε, ξεπερνούνται οι κόκκινες γραμμές του. Υπάρχουν λοιπόν προσπάθειες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στη διαδικασία και κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ή ακόμα και πριν από αυτόν μια συμφωνία. Προσπαθεί λοιπόν μέσω ψηφισμάτων εγκαίρως, ακόμα και πριν συντάξει η Κομισιόν τις ε, σχετικές οδηγίες, σχετική νομοθεσία, να δηλώνει την άποψή του. Μετά υπάρχει και η άτυπη ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις ε, διαπραγματεύσεις. Εδώ έχει ισχυρότερη θέση το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας και μαζί με αυτό της Νέας Ζηλανδίας, η οποία δεν ε, συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη. Τώρα, στις Ηνωμένε Πολιτείες τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχει πιο σημαντικό ρόλο το Κογκρέσο, διότι εάν ο πρόεδρος θέλει να κάνει κάτι, θέλει να συνάψει μια συμφωνία, μπορεί μεν να το κάνει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου, όμως ε, έχει περιορισμένες δυνατότητες. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τον Ιούλιο του 2021 όπου ο πρόεδρος μπορεί να υπογράψει μια συμφωνία χωρίς την έγκριση του Κοινοβουλίου, του Κογκρέσου. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει την συνταγματική αρμοδιότητα να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις. και είναι εκείνο που θέτει τους στόχους για τις ε, διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα και που θα λαμβάνουν χώρα τα επόμενα χρόνια. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι υπάρχει ένα Συμβούλιο Υπουργών, υπάρχουν πολλές φωνές, υπάρχει Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η διαπραγματευτική εντολή είναι και αυτή αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών. Το αποτέλεσμα είναι ότι το, η διαπραγματευτική αυτή διαδικασία μεταξύ ε, Συμβουλίου Υπουργών και Κοινοβουλίου οδηγεί σε πιο ε, καλά οριοθετημένους στόχους. Αυτά ως προς το στάδιο της εντολής. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών ο επικεφαλής διαπραγμάτευσης έχει λευκή επιταγή και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Σε καμία περίπτωση δεν συμβαίνει αυτό. Όταν ο πρόεδρος τον είπα θέλει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, πρέπει προηγουμένως να διαβουλευτεί με τις ειδικέ επιτροπές του Κογκρέσου για τους στόχους που θέλει να επιτύχει και για την για το κατά πόσο η συμφωνία που θέλει να επιτύχει συμφωνεί με τους στόχους της σχετικής ε, νομοθεσίας για την προώθηση του εμπορίου. Περνάμε τώρα στο στάδιο της διαπραγμάτευσης. Εδώ τα πράγματα είναι παρόμοια με το προηγούμενο στάδιο. Βλέπουμε ότι το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σίγουρα ισχυρότεροι και έχουν ισχυρότερη θέση ακριβώς διότι αμφότεροι κατανοούν ότι χρειάζεται να τεθεί σε ισχύ νομοθεσία. Ως αποτέλεσμα, και τα δύο όργανα μπορούν να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις, διαπιστεύονται καταλήλως, ενημερώνονται αμέσως και πλήρως για την πρόοδο των ε, διαπραγματεύσεων και για τις συνομιλίες. Και αυτό το στοιχείο της ενημέρωσης σημαίνει ότι υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν αλλαγές κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης. Στις Ηνωμένε Πολιτείε δηλαδή υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με αυτό που γίνεται εδώ, με τις συζητήσεις που γίνονται εδώ σε επιτροπές. Υπάρχει διαφορά όμως ε, με το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, διότι το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας δεν παίζει επίσημο ρόλο ε, στην ολοκλήρωση μιας συμφωνίας, Παρομοίω και ο Καναδά. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις του Καναδά και της Αυστραλίας μπορούν ε, να παρακάμψουν τα κοινοβούλια αν θέλουν να ολοκληρώσουν μια συμφωνία. Κάτι που δεν συμβαίνει ούτε εδώ ούτε στη ΣΥΠΑ. Βλέπουμε βέβαια, λέω και συχνότερα, ότι στις εμπορικές διαπραγματεύσεις υπάρχουν τεχνικά μέτρα τα οποία γίνονται όλο ένα και σημαντικότερα. Όχι γιατί οι συμφωνίες είναι κατά ανάγκη τεχνικές, αλλά γιατί οι εμπορικές συμφωνίες αφορούν και θέματα τα οποία έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνουν ομοθετικές ρυθμίσεις διασυνοριακά. Υπάρχει λοιπόν ένας καταμερισμός των αρμοδιοτήτων τόσο εδώ όσο και στο Κογκρέσο. Εδώ το βλέπετε με τις ομάδες παρακολούθησης, με τις συνεδριάσεις των επιτροπών, με τις ακροάσεις κτλ. Με τα ψηφίσματα που ε, εγκρίνει το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με την πρόσβαση στα έγγραφα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε λαμβάνει χώρα η ίδια συζήτηση από το 2007 με την κυβέρνηση Bush κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Νότια Κορέα, με τη Νότια Κορέα και με διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής είχε γίνει το ίδιο. Είχε ζητηθεί να αποκτήσει το Κοινοβούλιο περισσότερη πρόσβαση σε έγγραφα. Έτσι ώστε να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Και εγκρίθηκαν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά από το Αμερικανικό Κογκρέσο για την αύξηση της ε, διαφάνειας και της πρόσβασης των μελών του στις διαπραγματεύσεις. Εδώ τώρα στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε μια συνοπτική εικόνα και φαίνεται η σημαντική διαφορά μεταξύ Κογκρέσου και Ευρωκοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπουμε ότι σε τελική ανάλυση μπορεί να υπερψηφίσει ή να καταψηφίσει μια πρόταση. Το ίδιο συμβαίνει και στο Αμερικανικό Κογκρέσο, δηλαδή όταν ε, μία εμπορική συμφωνία καλύπτεται από τη σχετική εμπορική νομοθεσία, τότε το Κογκρέσο μπορεί να την υπέρει κατά ψηφίση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όταν οι πολίτες κάνουν μεγάλες υποχωρήσεις μέσω των εκπροσώπων τους, τότε θέλουν να είναι σίγουροι ότι οι παραχωρήσεις αυτές δεν θα υποστούν αποδυνάμωση μέσω τροπολογιών. Το Κογκρέσο λοιπόν παίρνει πίσω το προνόμιο που είχε δώσει στον πρόεδρό του, δηλαδή την δυνατότητα τροποποίησης μιας εμπορικής συμφωνίας. Αυτό συμβαίνει με δύο τρόπους. Είτε το Κογκρέσο, η Γερουσία ή η Βουλή των Αντιπροσώπων μετά από διαβούλευση καταλήγει στο ότι ο πρόεδρος δεν σεβάστηκε ούτε το πεδίο εφαρμογή ούτε τη διαδικασία διαβούλευσης που όφιλε βάσει νόμου όπως έγινε τον Απρίλιο του 2008 όταν ο πρόεδρος είχε υπογράψει τη συμφωνία με την Κολομβία. Και είδαμε ότι μετά από ένα χρόνο δύσκολων συνομιλιών της κυβέρνησης Bush για τη συμφωνία με Κολομβία, Περού, Παναμά και Νότια Κορέα. Όταν έφτασε στο στάδιο του Κογκρέσου, ο πρόεδρος έπρεπε να σεβαστεί διάφορες προσθήκες. Στην ουσία λοιπόν, τι γίνεται, το Κογκρέσο, είτε η Ανωτικά το Βουλή, μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον πρόεδρο μεν να συνάψει μια συμφωνία, όμως μπορεί να κρίνει ότι επειδή ας πούμε δεν σεβάστηκε την νομοθεσία, παίρνουμε πίσω τη δυνατότητα που του είχαμε δώσει. Να συμφωνήσει χωρίς τροπολογίες. Έπειτα, το δεύτερο είναι αυτό που βλέπετε κάτω στην διαφάνεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα δοκιμαστικά, διοδοκιμαστικές συνεδριάσεις, διάφορες, ε, διάφορα τεστ. Όταν δηλαδή ένα νομοσχέδιο υποβάλλεται από τον πρόεδρο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, τότε ο χρόνος μετρά αντίστροφα. Δηλαδή, το Κογκρέσο πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 15 μέρες ας πούμε. Πρέπει δηλαδή να παραπεμφθεί το θέμα σε αρμόδιες επιτροπές, στη Γερουσία, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και μέσα σε 45 μέρες από την στιγμή αυτή πρέπει να ε, ψηφίσουν στην Ολομέλεια και μέσα σε 90 μέρες πρέπει και, το, και η Γερουσία και η Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν ε, για την πρόταση. Υπάρχει λοιπόν πολύ, πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα και έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν εντός αυτής της προθεσμίας ε, πώς θα κινηθούν. Εάν δεν έχουν επίσημα υποβάλει νομοσχέδιο σχετικά με την εφαρμογή, τότε υπάρχει ευκαιρία ανεπίσημα να τροποποιήσουν ένα νομοσχέδιο. Προτού αυτό υποβληθεί προς έγκριση στο Κογκρέσο. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Διότι αυτή είναι η στιγμή που τα μέλη του Κογκρέσου έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν, να τοποθετηθούν και να ζητήσουν επαναδιαπραγμάτευση σε ορισμένα σημεία τη συμφωνίας. Και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει ξανά και ξανά. Κοιτάξτε, ας πούμε, τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας. Ε, για το βόλιο κρέας, για τα φαρμακευτικά προϊόντα, για το χείριο κρέα για τα αυτοκίνητα, με τη συμφωνία ε, με την Κολομβία, α πούμε. Υπήρχαν άλλα θέματα. Και η συμφωνία USMCA τώρα, η οποία είναι ο διάδοχος της ναύτα, έχει κολλήσει σε θέματα επιβολής και ειδικών διατάξεων για το φαρμακευτικό κλάδο. Γιατί το τονίζω αυτό τόσο πολύ, διότι αυτή η διαδικασία αντισταθμίζει λίγο αυτό το μειονέκτημα με την υπερψήφιση ή την καταψήφιση ενός ε, νομοσχεδίου. Και αυτή η δυνατότητα υπερψήφιση καταψήφισης είναι σαν ε, πυρηνικό όπλο για το Κογκρέσο. Όταν, ας πούμε, έχεις διαπραγματευτεί με έναν εξωτερικό εταίρο και υποβάλλεις ε, το τελικό νομοσχέδιο προς έγκριση, ρισκάρεις πολλά. Ρισκάρεις το Κοινοβούλιο να καταψηφίσει τη συμφωνία. Και αυτό που θέλουν και οι δύο εταίροι είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ακριβώς γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει εγκαίρως και νωρί στις διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε να καταδείξει τι θέλει και τι δεν θέλει στο πλαίσιο της συμφωνίας. Όταν όμως ολοκληρωθεί μια συμφωνία, τότε θα ε, υποβληθεί προς ε, υπέρ ή κατά ψήφιση σε τελικό στάδιο. Και στις ΗΠΑ εκεί μπορεί να καταποντιστεί μια συμφωνία. Για να το αποφύγουμε λοιπόν αυτό, αυτό το αδιέξοδο, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και η μέση Δηλαδή αυτά που λένε, αυτές που λένε οι τύποι, τύπου συνεδριάσεις, η, η άτυπη διαβούλευση Και έρχομαι τώρα στο συμπέρασμα. Γιατί διαπιστώνω ότι καταχράστηκε και λίγο το χρόνο. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά ήταν πολλά τα στοιχεία που ήθελα να σας δώσω. Λοιπόν, ποια είναι το συμπέρασμα. Και ποια είναι τα μηνύματα που θα ήθελα σήμερα να σας περάσω. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, γνωρίζει κανείς, να έχει την εξειδικευμένη γνώση σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε καταστάσει όπω τώρα που θα έχουμε τι ευρωεκλογέ που θα υπάρξει ανανέωση των ευρωβουλευτών. Οι συμφωνίε αυτέ είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει ότι όσοι διαπραγματεύονται, συζητούν για αυτέ, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τα τεχνικά θέματα. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν βουλευτή, ο οποίο έχει πολύ φορτωμένο πρόγραμμα ήδη. Γι' αυτό, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναπτύξει τη δική του, ε, το δικό του θεσμικό σύστημα για να κρατάει τη γνώση στο εσωτερικό του, πέρα από το πολιτικό προσωπικό δηλαδή. Και διευκρινίζω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο προσωπικό έτσι, ενδιαφέρον να προωθήσω τη γραφειοκρατία ή, να, ή το προσωπικό αλλά χρειάζεται με κάποιο τρόπο να κρατιέται αυτή η γνώση. Το δεύτερο είναι υπάρχει καλή και στενή συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα που έχουν την εμπειρία των διαπραγματεύσεων, δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα κράτη-μέλη. Στο γενικότερο πολιτικό παίγνιο το ευρωπαϊκό, ο μόνος παίκτη ο οποίος δεν έχει από πίσω του μια μεγάλη γραφειοκρατία να το υποστηρίζει, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίω υπάρχει κάποιο προσωπικό εδώ και υπάρχει υποστήριξη, αλλά αν συγκρίνεται το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το αντίστοιχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με τι δημόσιε διοικήσει των κρατών μελών, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση. Το δεύτερο ε, είναι κάτι το οποίο μα εξέπληξε. Είναι το γεγονό ότι σιγά σιγά κάποιες πρακτικές θεσμοποιούνται. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, συμβαίνει συχνά σε κοινοβουλευτικούς, στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο να δημιουργούνται τέτοιες παραδόσεις και κάποιες ε, ε, ανεπίσημες διαδικασίες όταν το ζήτημα είναι πολιτικό και όταν είναι ευαίσθητο. Ε, με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται οι ανεπίσημες διαδικασίες για να αντιμετωπιστούν ζητήματα τα οποία μπορεί να μην είναι ευαίσθητα ή επίμαχα μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά μπορεί να γίνουν αργότερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τι αξιοποιεί σε αυτέ. Και το τρίτο, δεν θα μπω και περισσότερο, σε περισσότερε λεπτομέρειε αυτό. Το τρίτο είναι όλα αυτά που σα είπα για την εφαρμογή. Επαναλαμβάνω λοιπόν αυτό που είπα και στην αρχή. Εάν ήμουν μέλο του Αυστραλιανού ή του Καναδέζικου Κοινοβουλίου θα ζήλευα το Ευρωπαϊκό γνωρίζουμε ότι πολλά μέλη αυτών των δύο κοινοβουλίων ε, κοιτούν και προσπαθούν να δουν ποιες πρακτικές έχει αναπτύξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο των Υπουργών για να τις αξιοποιήσουν ως εμπειρία και να ε, ενισχύσουν το ρόλο τους στις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Εάν ήμουν μέλος του Κογκρέσου θα ήμουν περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα και πώ θα αναπτύξει και την τεχνική του ικανότητα να παρακολουθεί τέτοιε δύσκολε διαπραγματεύσει. Και τρίτον, εάν ήμουν μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήμουν ευτυχή για αυτό που έχω σήμερα, αλλά θα πρόσεχα. Και θα προσπαθούσα να εντάξω σε επίσημε θεσμικές διαδικασίε πράγματα τα οποία σήμερα γίνονται ε, ανεπισήμω. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων στο μέλλον. Προεδρό, σα ευχαριστούμε. Για την ανάλυση που μας κάνατε και που μας εξηγείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι περήφανο και χαρούμενο για τις δυνατότητες που έχει. Πριν να δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους, θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα τη Βρετανή συνάδελφο που μετά τις 29 Μαρτίου βρίσκεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας τους καλωσορίζω όλους. Εγώ θα ήθελα να μπορούσα να τους καλωσορίσω για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι Λοιπόν, ποιο θέλει το λόγο για ερωτήσει. Ευχαριστώ στο συγγνώμη που δεν ήμουν από την αρχή της παρουσίασής σας. Σας ευχαριστώ για αυτό που είπατε, κύριε Πρόεδρε. Έχω πάθει μπρεξιτίτιδα, που είναι μια ασθένεια που προκαλεί αυτή η τραγική κατάσταση στη χώρα μου. Μέσω όμως της διαδικασίας του Brexit έγινε πολλή συζήτηση στο Κοινοβούλιο στην τη Βουλή των Κοινοτήτων για το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η εμπορική μας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήθηκε πάρα πολύ για το πώς λειτουργούν οι εμπορικές συμφωνίες και το εμπόριο γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση και η διαδικασία ήταν ενδιαφέρουσα. Γιατί με έκανε να σκεφτώ και πώς λειτουργούμε εμείς οι Βρετανοί ευρωβουλευτές. Δεν ξέρω πόσοι από τους συναδέλφου από άλλε χώρες είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα εθνικά του κοινοβούλια και να του εξηγήσουν στου συναδέλφους του, στι χώρε του, τι σημαίνει ακριβώ να είναι κανεί μέλος σε μια Επιτροπή διεθνού Εμπορίου, τι σημαίνει να έχει πρόσβαση σε έγγραφα, τι σημαίνει να έχει τη δυνατότητα να ανταλλάσσει απόψει επισήμω ή ανεπισήμω με αυτού που κάνουν τι διαπραγματεύσει. Ε, και συμφωνώ πλήρω με αυτό που είπατε, ε, ότι και το είδα και στην πρακτική μου εμπειρία παρακολουθώντας τις εμπορικές συμφωνίες και την πολιτική της Ένωσης ε, τα τελευταία 15 χρόνια. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας ότι η μεγάλη πρόοδος σημειώθηκε μετά από μεγάλα ζητήματα που ήταν ε, πολιτικά επίμαχα, ε, δημιούργησαν διαμάχες, όπως για παράδειγμα η TTIP. Υπήρξαν συγκρούσεις οι οποίες άρνηξαν δρόμος ή από την άλλη μπορεί να δίνεται πλέον λιγότερη σημασία σε ζητήματα τα οποία να, είναι, να μην είναι τόσο ευαίσθητα πολιτικά ή να είναι λιγότερο ενδιαφέροντα. Το ερώτημα λοιπόν που έχω ε, εγώ είναι πώς μπορεί κανείς να θεσμοποιήσει τις ανεπίσημες διαδικασίες χωρίς να, χωρίς να δημιουργήσει αγγυλώσεις, χωρίς να γίνουν πολύ ε, Γιατί χρειάζεται και μια κάποια ευελιξία η ανεπίσημη δυνατότητα παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντική, γιατί εδώ που τα λέμε η επίσημη δυνατότητα που έχει το Κοινοβούλιο είναι απλώ να απορρίψει, να εγκρίνει, να δώσει συγκατάθεση. Ε, ε μια διαδική επιλογή. Ενώ εγώ πιστεύω ότι η ευελιξία είναι πολύ σημαντική. Το δεύτερο. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα μας αποσχολεί όλο και περισσότερο και μάλιστα σήμερα στην ε, κυκλισμένων του θυρών συνεδρίασή μα για την Νότια και Κορέα θα συζητήσουμε, είναι ακριβώς το πώ το Κοινοβούλιο μπορεί να παρακολουθεί την εφαρμογή μια συμφωνίας μετά την επικύρωσή τη. Και ιδιαίτερα σε ζητήματα τα οποία είναι επιμαχά. Όπω για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευθύνη των επιχειρήσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα. Πώ μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι αυτέ οι διατάξει τι οποίε συμφωνήσαμε εφαρμόζονται όντω στην πράξη. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε εσείς και για αυτό το θέμα, για το ζήτημα τη εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ζητάει κανεί άλλο το λόγο. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φυσικά, θα ήθελα να θέσω και εγώ δύο ερωτήματα. Το ένα μοιάζει με την πρώτη ερώτηση για τις άτυπες δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θυμάμαι πολύ καλά στις διαπραγματεύσεις για τη ΣΥΤΑ και ειδικότερα για τη διαδικασία μετά από τη σύναψη της συμφωνίας αυτής με τον Καναδά. Τότε το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι με το παλιότερο σύστημα δεν θα είχε δεχθεί σε καμία περίπτωση το σύστημα, τη συμφωνία με τον Καναδά τη Συμφωνία ΣΥΤΑ και ακόμα και μετά από την ολοκλήρωση τη συμφωνία και τη σύναψή τη και το τέλο των διαπραγματεύσεων ε, υπήρχε δυνατότητα βάθρων αλλαγή του κομματιού για τι επενδύσει. Οπότε ποια είναι ε, αυτή η άτυπη δυνατότητα, αυτές οι άτυπες δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την εκτίμησή σας. Μπορούμε να αποφεύγουμε αυτές τις πυρηνικές όπως τις ονομάσατε λύσεις όπως μπορεί και το Κογκρέσο στη ΣΥΠΑ και τώρα για το Κογκρέσο φυσικά. Σαφώς ε, έχει ευθύνες το Κογκρέσο για την εμπορική πολιτική όπως θεσπίζεται στο Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. αλλά το γεγονό ότι με καταξιδότηση πράξη έδωσαν ε, στον πρόεδρο εξουσία για θέματα εθνικής ε, ασφάλειας το 232 το, και για το άλλο για την ε, αθέμητη συμπεριφορά εμπορικών εταίρων η εξουσία τελικά του Κογκρέσου είναι απεριόριστη ή περιορίζεται λόγω αυτών των, των αυτής της εκχώρησης εξουσιών στον πρόεδρο και τώρα ο Πίτερ Σέντερ από την Κομισιόν, ε, οι σχέσεις μας ε, ανέκαθεν ε, υπήρξαν σχηνοτενεί. Συχνά συζητούσαμε το πώ θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Θυμάμαι πολύ καλά, όταν ξεκίνησα εδώ ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, μόλις 23 μέλη του Κοινοβουλίου είχαν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, ενώ τώρα και τα 751 μέλη, όλα τα μέλη έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα εγγραφά. Συμφωνήσαμε να μην έχουμε προσωρινή εφαρμογή από την Κομισιόν πριν δοθεί η συνένεση του Κοινοβουλίου. Και συμφωνήσαμε και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Οπότε εξελίξεις ε, υπάρχουν και στις δυνατότητες ε, εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Μπέντ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μου δίνεις τη δυνατότητα να σχολιάσω αυτή την ενδιαφέρουσα έκθεση του καθηγητή Κέρμαντς. δίνει μια πολύ καλή εικόνα στις τρεις προτάσεις μας έδωσε για τις ε, τρεις θέσεις των ε, τριών κοινοβουλίων. Κάτι που αντιλαμβανόμαστε μέσα από αυτή την παρουσίαση, την έκθεση αυτή, είναι ότι στο επίκεντρο τη σχέση που καταφέρουμε να χτίσουμε την τελευταία πενταετία μετά από τη θέση ισχύ ειδικότερα τη συνθήκη Λισαβόνα, υπήρξε η σαφή ε, κατανόηση από μέρου τη Κομισιόν ότι σε τελική ανάλυση για να παίξει το Κοινοβούλιο το ρόλο του στην έγκριση και συνένεση στι εμπορικέ συμφωνίε πρέπει να εμπλέκεται πολύ στενά και να ενημερώνεται πλήρω σε ολόκληρη τη διαδικασία της προετοιμασίας και της ε, πραγματοποίησης των ε, διαπραγματεύσεων. Όχι μόνο νομικά είναι σωστό δυναμή των υποχρεώσεων μας ε, όπως τις προβλέπει η συνθήκη, αλλά είναι και το σωστό να γίνεται αυτό. Υπό αυτό το πνεύμα, μάλιστα, η Κομισιόν έχει προσεγγίσει τη σχέση αυτή, προσπαθώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό να παρέχει πλήρες πληροφορίες αναφέρατε στην πρόοδο που έχει γίνει, ειδικότερα όσον αφορά την πρόσβαση στην έγγραφα αυτά καθεαυτά. Κοιτώντα την τελευταία πενταετία και τα σχετικά νούμερα, πάνω από 1.700 έγγραφα έχουμε μοιραστεί με την Επιτροπή ΙΝΤΑ εδώ του Κοινοβουλίου. Έχουμε απαντήσει σε 1.600 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και στο πλαίσιο αυτών έχουμε και δημιουργικούς ευέλικτους μηχανισμούς όπως ομάδες παρακολούθησης ή τεχνικές συνεδριάσεις που θεσπίστηκαν ε, με στόχο την εμβάθυνση της αλληλοσυνεννόησης και της συνεργασίας με την Επιτροπή σας, ε, ώστε να έχει τη δυνατότητα να διδραματίσει το ρόλο που της αρμόζει. Και αυτή η ευελιξία, πιστεύω, βρίσκεται στο επίκεντρο της σχέσης μας. Αυτό αναγνωρίζεται και στην έκθεση. Η έκθεση επισημαίνει πολύ καλά, πιστεύω, τις δυσκολίες που θα έχει να αντιμετωπίσει το νέο κοινοβούλιο. Συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη θεσμική μνήμη ε, στο Κοινοβούλιο και τη διατήρησή της. Η τεχνική προγνωμοσύνη είδαμε μια μελέτη, ε, είδαμε ότι ε, αυξάνεται η συμμετοχή στις μελέτες σε αυτή την Επιτροπή και αυτό είναι από τα δύσκολα σημεία για τη νέα Επιτροπή που θα συσταθεί, αλλά υπάρχουν οι σωστές ομάδες για να ε, σας προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη. Φυσικά, όσον αφορά τους άτυπους μηχανισμούς ε, ε, που λειτουργούν καλά, πρέπει να κινούμαστε εντός των περιθωρίων που προβλέπει η συνθήκη και για η κωδικοποίηση των άτυπων μηχανισμών, όπως αναφέρατε και εσείς, μπορεί μερικές φορές να αποδείχνεται δύσκολη. Όταν απαιτούνται λύσεις οι οποίε πρέπει να δοθούν γρήγορα. Αλλά πιστεύω ότι μετά από την συνθήκη τη Λισαβόνα και την εκλογή αυτού του τελευταίου κοινοβουλίου, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο συνεργάστηκαν πολύ στενά και πολύ καλά για να σημειωθεί προ, κάποια πρόοδο. Πιστεύω λοιπόν ότι στην εκθέση αναφέρονται πολύ καλά κάποιε από τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Παρουσιάζονται κάποια στοιχεία προ προβληματισμό καθώ περνάμε στο επόμενο κοινοβούλιο και θα πρέπει να ξέρετε ότι και στο επόμενο κοινοβούλιο η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται ανοιχτά και διαφανώς. Και θα υποστηρίζει το Κοινοβούλιο σε να διαδραματίσει τον πλήρη ρόλο του στην ανάπτυξη και στι εξελίξει τη εμπορική πολιτική. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, μπορώ να σα διασφαλίσω ότι ναι, θα διαδραματίσει το Κοινοβούλιο αυτό το ρόλο. Ωραία, λοιπόν. Ε, κύριε Κέρμαν, παρακαλώ. Okay. Θα ήθελα να ξεκινήσω για την, λέγοντας για την εφαρμογή. Όταν εξετάζουμε την εφαρμογή μιας εμπορικής συμφωνίας, σίγουρα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πιο αδύναμος η περίπτωση των ΙΠΑ είναι συγκρίσιμη θα έλεγα, διότι στο Κογκρέσο είναι πολύ προσεκτική σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων μιας συμφωνίας, διότι έχουν επίγνωση του ότι από τη στιγμή που συναυθεί μια συμφωνία χάνουν μέρος του ελέγχου τους. Αν δείτε τι έγινε στην περίπτωση της συμφωνίας με το Περού και με τη Γουατεμάλα, αλλά και σε όλη τη συζήτηση με την ε, Κολομβία και τα προβλήματα με τα εργασιακά δικαιώματα. Και επίσης τις συζητήσεις για τη νέα συμφωνία USMCA και τα περιβαλλοντικά και εργασιακά ζητήματα, θα δείτε ότι το Κογκρέσο έχει αυξημένη ευαισθησία για τα θέματα αυτά, ακριβώ διότι συνειδητοποιεί ότι από τη στιγμή που συναυτεί μια συμφωνία πρέπει και να εφαρμοστεί. Και αυτό είναι το σημείο όπου χάνει τον έλεγχο. Και ε, η ερώτηση του Προέδρου για τα 232 και 231 και 301. Αυτά είναι παραδείγματα μέτρων που ελήφθησαν από τον εκτελεστικό κλάδο της εξουσίας. Και αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ υπάρχουν δύο νομοσχέδια υποσυζήτηση, τα οποία βέβαια απέχουν πολύ από το να βρουν πλειοψηφία που να τα εγκρίνει. Όταν ο πρόεδρος λαμβάνει μέτρα υπό το 232, το κάνει γιατί αυτά είναι περιοριστικά εμπορικά μέτρα που έχουν βάση στην εθνική ασφάλεια. Όπως για παράδειγμα ό,τι έγινε στην περίπτωση του Χάλβα και της αυτοκινητοβιομηχανίας το 1962. Το Κογκρέσο όταν πρέπει να εγκρίνει ένα μέτρο που έχει λάβει ο πρόεδρος ε, σύμφωνα με το άρθρο 232, η προθεσμία είναι 75 ημέρες. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το Κογκρέσο μπορεί να μην εγκρίνει τα μέτρα που λαμβάνει ο πρόεδρος και εδώ πρέπει να βρει την πλειοψηφία να το κάνει. Αν δεν έχει πλειοψηφία τότε τα μέτρα περνάνε, ό,τι και να γίνει. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να δούμε τις σχέσεις ε, μεταξύ του Κογκρέσου και του Πρόεδρου. Είναι πολύ δύσκολο Μέλο του Κογκρέσου να αμφισβητήσει την εξουσία του Προέδρου σε θέματα εθνική ασφάλεια. Υπάρχουν όμως διάφορα άλλα μέτρα όπου μπορείτε να φανταστείτε ε, πως συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί οι σχέσεις δεν είναι τόσο αυστηρά ιεραρχημένες. Και εκεί το Κογκρέσο μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του Προέδρου σε αντίθεση με θέματα εθνική ασφάλεια. Τώρα, στην περίπτωση της συμφωνίας ΣΥΤΑ, αν δεν κάνω λάθος, είναι μια περίπτωση όπου φαίνεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου κατά την προετοιμασία μιας διεθνούς συμφωνίας. Βέβαια, υπάρχουν και οι κίνδυνοι. Για παράδειγμα, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν φροντίσει να συμμετάσχει ενεργά στη διαδικασία, στις διαπραγματεύσεις συμφωνιών, οι οποίες είναι αρκετά αμφιλεγόμενες, μπορεί να έχει αυτό απρόβλεπτα αποτελέσματα για τους ε, διαπραγματευτές της Κομισιόν. Και γιατί αυτό, διότι ξαφνικά βλέπουμε να κινητοποιείται η κοινωνία και να εμφανίζονται θέματα που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια ξαφνικά, θέματα τα οποία είναι αρκετά ε, σημαντικά για τους πολίτες και αυτό έγινε στην περίπτωση της Συμφωνίας ΣΕΤΑ. Υπήρξε ένα έντονο κίνημα πολιτών, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Κύριε καθηγητά, διακόπτει πρόεδρο, δεν θέλω να σα διορθώσω, όμω το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ψηφίσει ένα σχετικό ψήφισμα για τη συμφωνία ΣΥΤΑ πολύ πριν γίνουν όλα αυτά που λέτε πολύ πριν την κινητοποίηση, πολύ πριν ζητήσουν οι πολίτε εξυγχρονισμό του συστήματο κτλ. Ναι, ναι, με συγχωρείτε. Ε, Όπω σα είπα και πριν, ε, δεν είμαι μέσα για να τα γνωρίζω. Εξωτερικό παρατηρητή είμαι. Αλλά ας δούμε για παράδειγμα τις ε, συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ είναι μια περίπτωση ενδεικτική. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει έναν αξιόπιστο εταίρεο έτσι ώστε να μην αβαγίσουν οι διαπραγματεύσεις, έτσι ώστε αν ε, φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πει εντάξει εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε αλλά αφού δεν γίνεται αλλιώς θα εγκρίνουμε τη συμφωνία. Τέλεια, υπέροχα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε και σας ευχαριστούμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 6. Πουλερικά. Κρέας πουλερικών και το σχέδιο συμφωνίας για τροποποίηση του δασμολογικού καθεστώτος στη συμφωνία με την Ουκρανία. Έχουμε εκπροσώπους ε, της Κομισιόν εδώ. Υπάρχει πρόταση να αλλά... η πρόταση από την Κομισιόν να αλλάξει η Συμφωνία Σύνδεσης για την ε, αλλαγή κατηγορίας στις εισαγωγές ε, κρέας πουλερικών. Πρόκειται για μια συμφωνία η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή προσωρινά και λάβαμε μια επιστολή από τους επιτρόπους Μάλμστρομ και Χόγκαν, οι οποίοι μας ζητούν να δεχτούμε την αρχική συμφωνία, προτού το Κοινοβούλιο δώσει και επίσημα τη συγκατάθεσή του. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Σάιφη, η οποία αντικαθιστά την κυρία Χούμπνερ, η συγγήτρια, και τον κύριο Βαλέσα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο κύριος Βαλέσα δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίασή μας σήμερα για λόγους οικογενειακού, Ζητά συγγνώμη και θα διαβάσω την παρέμβασή του. Ως τακτικός συζητητή για την Ουκρανία, ο κύριο Βαλέσα παρακολουθεί την κατάσταση της χώρας, όχι μόνο όσον αφορά το εξωτερικό τη εμπόριο, αλλά κυρίω όσον αφορά την πολιτική κατάσταση. Η Ουκρανία έχει λάβει μέτρα φιλελευθερωποίηση και ειδικά μέτρα για, τους, για, για το τελευταίο καθεστώ, για του δασμούς. Τα πουλερικά, με, σε, επί τη βάση τη συμφωνία, έχουν ειδικό δασμολογικό καθεστώς. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι είχε ε, αυξηθεί η εισαγωγή πουλερικών από την ε, Ουκρανία, ιδιαίτερα αυτό ε, εξαιτία του δεσμολογικού καθεστώτος το, η συμφωνία δεν προέβλεπε κάποιο ποσοτικό όριο. Αυτή η μεγάλη αύξηση μεταφράστηκε σε μια αύξηση από 3.700 ε, τόνους το 2016 σε 55.000 τόνους το 2018. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινητοποιήθηκε το ζήτημα αυτό την προηγούμενη άνοιξη, το ερεύνησε και επιβεβαιώθηκε ότι αυτό που γίνεται από τις εισαγωγές είναι να χρησιμοποιούν ένα δασμολογικό καθεστώς μηδενικό, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει, δεν αντιστοιχεί στη σωστή περιγραφή του εμπορεύματο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταφέρουν να εισάγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολερικά σε πολύ μεγάλες ποσότητες και χωρίς δασμούς. Θεωρούμε ότι μια και θεωρήσαμε λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία είναι απαράδεκτη, χρησιμοποιήθηκε οι σχετικές προβλέψεις της ε, DCFTA, της ε, συμφωνίας. Το επισημαίνει και αυτό ο κύριος Βουβαλέσα και ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση της Ουκρανίας για να λεφθεί το ζήτημα αυτό. Βέβαια αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο ε, περίπλοκη για την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τις προεδρικές εκλογές Και αυτό των λεχθέντων, ο κύριος Βαλέσσα ζητά να ε, επικυρωθεί αυτή η συμφωνία από την Ουκρανία και να δώσουμε την εγκρισή μας για την εφαρμογή της, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η εισαγωγή πουλερικού από... χωρίς έλεγχο. Ο κ. Βαλέσα συμπληρώνει ότι έχουμε καθήκον ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προσπίσουμε τους Ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Συμφωνώ πλήρω, κύριε Πρόεδρε, με αυτή την δήλωση του κύριου Βαλέσα ως υπεύθυνη για ζητήματα διεθνούς εμπορίου. Θα ήθελα να επισημάνω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει, έχει πο, πολλές φορές ζητήσει την Επιτροπή να παρεμβαίνει γρήγορα όταν υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Τα πουλερικά δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται με τέτοιον τρόπο είναι απαράδεκτο να δημιουργούνται προβλήματα στου Ευρωπαίου κτηνοτρόφου εξαιτία αυτή τη λειτουργία στην συμφωνία. Θα πρέπει λοιπόν να, να δράσει, να ληφθούν μέτρα για τον έλεγχο των εισαγόμενων προϊόντων και για τον σεβασμό των ποσοτικών ορίων που έχουμε συμφωνήσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στο, στον συνάδελφο, όχι δεν είναι εδώ ο συνάδελφο ο πρόεδρο τη Επιτροπή. Αγροτικής ανάπτυξη. Άγκρι, είστε εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πήρα την ευκαιρία λοιπόν για να τοποθετηθώ και εγώ στη συζήτηση αυτή, διότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ο τομέας λοιπόν των πουλερικών και οι εισαγωγές πουλερικών, κρέατος πουλερικών από την Ουκρανία προκαλούν προβλήματα στην εσωτερική αγορά. Φυσικά και κατανοούμε τη θέση της Ουκρανίας και θέλουμε να βοηθήσουμε τη χώρα και τους αγρότες της, τους πραγματικούς αγρότες Δεν μπορούμε όμως να δεχτούμε αυτά τα παραθυράκια και την εκμετάλλευση που συμβαίνει. Διότι αυτή τη στιγμή πρόκειται περί εξαπάτησης Και βέβαια αναγνωρίζω το ότι οι διαπραγματεύσεις κρατάνε πάρα πολύ ακριβώς διότι δεν ήταν δυνατόν να έχουμε προβλέψει τα πάντα από πριν. Σχετικά με, τους, ε, με την ε, μηδενική δασμολογική κλάση, Αυτή η πρακτική λοιπόν ε, που βλέπουμε σε εισαγωγές από την Ουκρανία ότι κόβουν το κρέας με τρόπο που το χαρακτηρίζουν ε, ως άλλα τεμάχια και το πουλάνε ως στήθος κοτόπουλου είναι αθέμητη. Είναι εις βάρος των δικών μας κτηνοτρόφων και φυσικά ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι ανοιχτή προς την Ουκρανία, να ανοίξει και τις αγορές της για τα προϊόντα από την Ουκρανία, όμως η πρακτική ε, της Ουκρανίας ε, συνιστά ανήθικη εκμετάλλευση. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία ε, εκμεταλλεύτηκαν. Οφείλουμε λοιπόν να τηρούμε ορισμένες αρχές και τώρα και στο μέλλον. Η Ουκρανία είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλες δυνατότητες έχει έφορο έδαφος, καλό κλίμα και οι πρακτικές αυτές ε, μπορεί να οδηγήσουν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός, ε, εις βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις βάρος των δικών μας κτηνοτρόφων, όχι μόνο κτηνοτρόφων, αλλά και αγροτών. Υπάρχουν διάφορα ε, φρούτα, σμέουρα, φράουλες κτλ. Και είχαμε προβλήματα από την Ουκρανία στην Ανατολική Πολωνία, Όμω δεν είμαστε οι μόνοι. Του χρόνου μπορεί να έχει προβλήματα η Τσεχία, η Σλοβακία με τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία. Τώρα, διαπραγματευτήκαμε και άλλες συμφωνίες και τη συμφωνία με τον Καναδά Και παρατηρώ ότι δεν είναι μόνο η Ουκρανία δυνάμει επικίνδυνη, υπάρχουν και άλλε χώρε. Όμω στην περίπτωση τη Ουκρανία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα τα πράγματα ακριβώ επειδή έχει μεγάλη παραγωγή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το εμπάργκο στη Ρωσία οδήγησε στη Ρωσία να εξάγει χείριο κρέας σε μεγάλες ποσότητες σε τρίτες χώρες. Τώρα στα οποροκυπευτικά είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. και έτσι η παραγωγή ε, μεταφέρθηκε στη Ρωσία. Αυτή η κατάσταση λοιπόν ε, ε, βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΙΝΤΑ για την υποστήριξή της και που έδειξε βούληση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Αλλά αυτό σχετίζεται με ορισμένες παραχωρήσεις που έχουμε προσφέρει εμείς όσον αφορά τις ποσότητες, τις ποσοστώσεις που έχουμε παραχωρήσει στην Ουκρανία. Και αυτό επηρεάζει σημαντικά τη δική μας αγορά. Μην εκπλήσεστε λοιπόν αν ξαφνικά οι ε, γεωργοί μας ε, επικρίνουν. Αν δεν υπάρχει κάποια αναλογικότητα, εάν δεν τηρούνται οι αρχές της ανταγωνιστικότητας που επικρατούν στη δική μας ενία αγορά, όπως συμβαίνει εδώ, ε, σήμερα ουσιαστικά έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην αγορά γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη. Η επιρροή είναι μεγαλύτερη, ε, περισσότερα η επιρροή έχουν οι δραστηριότητες τρίτων χωρών παρά η ίδια η ΚΑΠ. Οπότε εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να δράσουμε και να παρακολουθούμε την αγορά αυτή και μέσω των δικών μας επαφών ε, που έχουμε απευθείας με τους παραγωγούς και γεωργούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σκιώδης ε, για τους σοσιαλιστές ε, δεν βρίσκεται εδώ. Μου έδωσε κάποιες σημειώσεις. Φυσικά ζητά συγγνώμη που δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ. Υποστηρίζει τη θέση του εισηγητή και έχει δύο ερωτήσεις. Στην πρόταση της Κομισιόν στην απόφαση υπάρχει μια συνολική αύξηση του ποσότητα διαρκείου και ο κ. θέλει να μάθει πώ αυτό επηρεάζει, αυτή η τροπολογία, πώ θα επηρεάσει τα πράγματα. Και δεύτερον, όσον αφορά την εξήγηση των κανόνων καταγωγής, ο κύριος Γκαμπλίκ κατάλαβε ότι δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή ή η καταγωγή των πολερικών όταν αφαιρείται το κομμάτι με το οστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να μάθει σε τι οφείλεται αυτό και τι αποτελέσματα, τι συνέπειες μπορεί να έχει. Τώρα για τους πρασίνους, ο κ. Μπάιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σπάνια έρχονται εδώ στην ίντα τα μέλη της Ευρωπίτροπης ε, Γεωργίας ε, όπως γνωρίζω. Αλλά έρχομαι σήμερα γιατί εδώ διακυβεύεται ο γεωργικό Τομέα Για άλλη μια φορά πάλι λόγω των συμφωνιών ελευθερών και θα πέρασω στα γερμανικά για τους μεταφραστές. Θα, κάνει λίγο, θα μου διευκολύνει την κατάσταση. Λοιπόν, συνοψίζω. Μιλάμε για μια εταιρεία που λέγεται MHP και η οποία παράγει πάνω από 1.200 τόνους κρέατος πουλερικών ετησίων που προμηθεύει 40% της αγοράς στην Ουκρανία και της οποίας ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε δισεκατομμύρια και που ε, διαφεύγει της φορολογίας. Ε, δεν θα δηλαδή εδώ στην Ουκρανία. Μιλάμε για μια πολυεθνική που μεγιστοποιεί τα κέρδη της, για να συνοψίσω. Οι ελεύθερες συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής ήταν 20.000 τόνοι ε, κρέατος πουλερικών που έφταναν στις αγορές μας με μηδενικό δασμό. Μιλάμε για στήθη κοτόπουλων, το καλύτερο κομμάτι δηλαδή του ζώου. Η επιχείρηση αυτή κατάφερε να βρει ένα παραθυράκι στην νομοθεσία και το εκμεταλλεύεται πλήρως. Δηλαδή συνειδητά, εσκεμμένα ε, παραμερίζει τους κανόνες αυτή η πολυεθνική φέρνοντας εδώ τα στήθη κοτόπουλου στην Ευρώπη με ένα μικρό κόκαλο ε, και έτσι δεν χρειάζεται να καταβάλει τις ποσοστώσεις, ε, τα ε, δασμούς που θα έπρεπε να καταβάλει. Και έτσι δεν τηρεί τους κανόνες. Επιπλέον, οι τελωνικές αρχές των κατοχωρών... χωρών ε, τόνισαν αυτό το πρόβλημα ήδη το 2017 και το 2018. Ήδη δηλαδή οι τελωνικές αρχές ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε ε, ενέκριναν τελικά αυτή την πρακτική. Τα τελωνία δηλαδή δέχθηκαν να μπουν στην Ευρώπη αυτά τα στήθη κοτόπουλου με το κοκαλάκι αυτό και ε, τα χαρακτήρισαν ως όχι στήθος κοτόπουλο, οπότε είχαν μηδενικά, μηδενικούς δασμούς και απαλλάχθηκαν από οποιοδήποτε δασμό. Η Προεδρία του Συμβουλίου έδωσε εντολή στην Κομισιόν για να επαναδιαπραγματευτεί το κεφάλαιο αυτό. Αυτό που θα με ενδιαφέρει, αγαπητή Επιτροπή, μπορείτε να μα πείτε αυτή την εντολή τι περιέχει. Η Κομισιόν μα το λέει πολύ καλά. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μιλάμε για πάνω από 50.000 τόνου εισαγωγών ετησίω. Μιλάμε για αύξηση 1000% εντό τριετία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι σημαντικό. Τι κάνει λοιπόν η Κομισιόν, ποια είναι η πρόταση τη Κομισιόν είναι να μας λέει τώρα, αφού έχουμε φτάσει στους 55.000 τόνους εισαγωγών, τι να κάνουμε, νομιμοποιούμε τις ποσότητες αυτές που εισήχθηκαν, που εισήχθησαν παράνομα στην Ευρώπη και μετά θα δώσουμε ποσόστοση επιπλέον 0%, με 0% ε, δασμούς και σε άλλα στήθη κοτόπουλου. Γιατί? Γιατί ξέρουμε ότι όλα τα κομμάτια του κοτόπουλου δεν υπόκεινται σε τέτοια δασμολογική ποσόστοση. Τι κάνουμε εδώ δηλαδή, παρακάμπτουμε την νομοθεσία. Στην αρχή είχαμε μιλήσει για 20.000 τόνους εισαγωγέ και με επιχορηγήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα βοηθήσαμε την αγορά τη Ουκρανία. και με επιχορηγήσει τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τελικά επιτρέψαμε σε αυτήν την επιχείρηση να αποκτήσει κυρίαρχη θέση στην Ουκρανική αγορά. Εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν εκεί ώστε αυτή η εταιρεία να εξαγοράσει μια εταιρεία μεταποίησης ε, κρέατος πουλερικών στην Σλοβενία όπου γίνεται αυτή η μετατροπή των, ε, ε, του στήθους αυτό που αναφέραμε, του στήθους Κοτόπουλου. Δώσαμε λοιπόν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα να δώσει και νέες πιστώσεις μάλιστα σε αυτή την επιχείρηση η οποία κατατρώει την Ουκρανική αγορά και σιγά σιγά θα δημιουργήσει προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή τα κομματιά αυτά κοτόπουλου, καρτιλίτερης ή χειρότερη ποιότητα, τελικά μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και θα του αναδώσουμε άλλε 50.000 τόνου ε, εισαγωγή κρέατο πουλερικών. Αυτό θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα για του δικού μα. Αγρότε. Δεν το χρειαζόμαστε οι Ουκρανοί παραγωγή. Δεν σέβονται του κανόνε που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο τη συμφωνία ε, που συμφωνήθηκε το 2013 και τότε ο κανόνα είχε ω εξή. Πρέπει να τηρούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο σε θέματα προστασία των ζώων. Ήδη τότε οι Ουκρανοί είχαν πει εμεί έχουμε ένα σχέδιο δράση που τρέχει μέχρι το 2017. Συγγνώμη, ένα σχέδιο δράση δεν είναι δράση. Ωραία, ακούγεται ένα σχέδιο, αλλά μπορεί να είναι ό,τι να είναι. Και μέχρι στιγμή το καν το έχουμε δει αυτό το σχέδιο δράση. Ούτε ξέρουμε αν τηρεί του ευρωπαϊκού κανόνε για την καλή μεταχείριση των ζώων και η Κομισιόν τη ΟΠΑ. Και σήμερα ξαφνικά εμφανίζεται μια πολυεθνική εταιρεία η οποία χρηματοδοτείται με ευρωπαϊκά χρήματα και κάνει αθέμητο ανταγωνισμό στον τομέα των πουλερικών, στην αγορά των πουλερικών στην Ευρώπη. Μα αυτό είναι γελίο, είναι καταστροφή για την ευρωπαϊκή παραγωγή. Θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να μα πει τι κάνει. Για να μην αναφερθώ στου κανόνε για την προστασία των ζώων και για την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτέ οι μηδενικών δασμών εισαγωγέ ξέρουμε ότι γίνονται χωρί σεβασμό των δικαιωμάτων των ζώων και επιπλέον του δίνεται και άλλη ποσόστοση και θα νομιμοποιήσετε και ότι εισήχθη στο παρελθόν παράνομα. Ειλικρινά, η Κομισιόν μας οφείλει εξηγήσει. Και ε, πέραν αυτού, παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο, ενώ έχετε την υποχρέωση να λάβετε την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίκυνται εκλογές. τι σα επηγητώ το, τόσο σήμερα που δεν μπορείτε να περιμένετε το επόμενο κοινοβούλιο. Ξέρω ότι στο Συμβούλιο τέλη του Μαΐου θέλετε να λάβετε αποφάσει, αλλά εγώ θα το παρακολουθώ στενά. Θα δω ποιο θα το ψηφίσει, Ποιο θέλει να παρακάμψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο εκμεταλλευόμενο την προεκλογική περίοδο. Και έτσι θα κάνω και θα το προσέξω και δεν θα σα αφήσω ήσυχου. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σόλτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν εξαιρετική η παρέμβαση του συναδέλφου που προσπαθεί να υπερασπιστεί από την πλευρά των σοσιαλιστών τον τομέα των πουλερικών, όμως είχαν υπερψηφίσει στους ελευτές, εάν δεν απατώμε αυτή τη συμφωνία με την Ουκρανία και είχαμε πει και το είχαμε επισημάνει και από τότε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ε, χρησιμοποιηθεί αυτή η συμφωνία για να υπονομευτούν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα έχουμε την απάντησή μας. Η MHP, ε, ε, η Ουκρανική, η οποία έχει κάνει μάλιστα και επενδύσεις στην περιοχή του Σουτρέχτης, αξιοποιεί ένα παραθυράκι για να περνάει με μηδενικούς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιες ποσότητες πουλερικών. Και με αυτές λοιπόν τις πρακτικές, τις οποίες καταγγέλουμε, έχουμε ε, που κρέας πουλερικών, πουλερικά να εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με, όχι μόνο με 0% δασμό, με, με μηδενικό δασμό, αλλά χωρίς να γνωρίζουμε και αν έχουν τηρηθεί οι κανόνες για την ασφάλεια, την διατροφική και την ευζοία των ζώων. Και αναρωτιέμαι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά. Μιλούμε για εξαγωγέ. ε, μεγάλο, σε μεγάλα επίπεδα, σε μεγάλες ποσότητες. Αυτή με αυτή την κατάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπονομεύει τον ε, τομέα των ε, κτηνοτρόφων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ενισχύει και ενθαρρύνει την εισαγωγή ε, πουλερικών τα οποία έχουν παραχθεί με συνθήκες πολύ χειρότερες. Και δημιουργεί αυτό προβλήματα σε πολλές χώρες. Μπορεί να αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δημιουργείται πρόβλημα του ανταγωνισμού και γιατί δεν λαμβάνουμε μέτρα για να καταπολεμήσουμε και να σταματήσει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός και να πιέσουμε, να, φροντίσουμε έτσι ώστε οι Ουκρανοί να σεβαστούν τη συμφωνία μας. Για το ΙΕΝΕΦ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους τους προλαλήσαντες και με το εμπάργκο στη Ρωσία γνωρίζουμε ότι οι κτηνοτρόφοι Ευρωπαίοι από το 2017 ήταν αυτοί που επλήγησαν με πρακτικές που γνωρίζουμε. Και έχει εξελιχθεί το φαινόμενο, όμως ότι αυτό που ήδη επισημάνθηκε και αυτό το οποίο πραγματικά εμένα με κάνει να ξανίσταμε είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να μας παρακάμψει και προσπαθεί να παρακάμψει και να παραγνωρίσει τις αρμοδιότητες που έχουμε για κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις αρμοδιότητες που έχουμε στο πλαίσιο του, του νομοθετικού ελέγχου. Ε, σήμερα μα ζητείτε να εγκρίνουμε κάτι το οποίο θα διευκολύνει του κτηνοτρόφους τη Ουκρανία. Όμω εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα μια απαράδεκτη πρακτική Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, η οποία παρεπιπτόντω να, να υπενθυμίσουμε ότι είχε υποστηρίξει τι κινητοποίησει στο Μαϊντάν και όλες τις αντίστοιχε πολιτικές ε, προεκτάσεις τους. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή, αυτή είναι μια πολιτική κίνηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντισταθεί. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό στην Επιτροπή. Είμαστε οι εκπρόσωποι δημοκρατικά εκλεγμένοι των Ευρωπαίων πολιτών και θα πρέπει να αντισταθούμε σε αυτή την επίθεση που γίνεται στι αρμοδιότητε μα και στι δυνατότητε μα από την πλευρά τη Επιτροπής. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε όλα αυτά να συμβαίνουν ε, και να παραμένουμε σιωπηλοί. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραγνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλά θέματα, όχι μόνο ε, στα αγροτικά, ε, γιατί στην πραγματικότητα δεν δέχεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό που εξασφαλίζει την δημοκρατία στην Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το... Θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα πριν δώσω το λόγο. Δεν είναι ξεκάθαρο τι θα σημάνει για τους Ευρωπαίους παραγωγούς αυτή, αυτό το, αυτή η ποσόστοση, αυτή η νέα ποσόστοση. Κατάγουμε, όπως ξέρετε, από την Γερμανία δεν παράγουμε μόνο αυτοκίνητα, έχουμε και ισχυρή αγροτική οικονομία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι θα οδηγήσει αυτή η αύξηση της ποσόστασης. Ο κύριος Πέτρος ε, Σουρμελής από την Γενική Διευθύνση Εμπορίου και η κυρία Σουζάνα Μάρσουέλα από την Γενική Διευθύνση Αγροτικής Ανάπτυξης από την Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο για το ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ επίγον και το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μιας και παρατηρούμε μια εκθετική αύξηση των εισαγωγών συγκεκριμένων ε, προϊόντων ε, πουλερικών από την Ουκρανία, όπως το ανέφεραν και συνάδελφοί σας. Αξιοποιώντας ε, μηδενικούς δασμούς, αναφέρθηκαν ήδη τα ποσά, από 3.700 τόνους το 2016, 55.000 τόνοι το 2018 την αύξηση. Είναι σημαντικό να τονίσει κανείς ότι εδώ δεν έχουμε ιστορικά δεδομένα για, και πρόκειται για δύο δεσμολογικές κατηγορίες οι οποίες με βάση την εμπορική, την FTA απελευθερώθηκαν. Τότε που έγιναν οι διαπραγματεύσει και συνήθιε αυτή η εμπορική συμφωνία, δεν θα μπορούσε κανεί να έχει προβλέψει ότι θα γίνουν τέτοιες ε, καταχρήσει των δασμολογικών ποσοστώσεων. Τότε δεν μπορούσε να το προβλέψει κανεί. Θα έχουμε λάβει επίσης από διάφορες τελωνιακές αρχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα δασμολόγια τους, και με βάση τα οποία προσπαθούν να φροντίζουν να γίνεται σωστά η κατηγοριοποίηση του εμπορεύματος, στη σωστή κατηγορία. Δεδομένου ότι για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ο δασμός είναι μηδενικός, δημιουργείται, ε, δημιουργούνται μεγάλες ανησυχίες και σε ενδιαφερόμενα μέρη και σε κράτη-μέλη ε, και φυσικά όπως είδαμε και σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε λάβει επιστολές πολλές που, που ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και να λύσει το πρόβλημα γρήγορα. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν σε αυτές τις ε, παρατηρήσεις, σημάνσεις που μας έγιναν, ξεκινήσαμε κάποιες διαρευνητικές συζητήσεις το 2018 με την Ουκρανία Καταθέσαμε μια πρόταση, ζητήσαμε εντολή διαπραγμάτευση τον Δεκέμβριο του 2018 για να διαπραγματευτούμε με την Ουκρανία μια περιορισμένη έκταση τροποποίηση τη FTA και οι διαπραγματεύσει αυτέ ολοκληρώθηκαν αρχέ Μαρτίου. Το λέω αυτό επίσης για να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει το ζήτημα ε, επιγόντως ε, και προσπαθήσαμε πάρα πολύ γρήγορα να υποβάλουμε την πρότασή μας στο Συμβούλιο για να μας δώσει πραγματευτική εντολή. Επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, μας έδωσε αυτή την εντολή μέσα σε ένα μήνα που σημαίνει ότι και το Συμβούλιο κατάλαβε πόσο επίγον είναι το θέμα. το προσχέδιο της συμφωνίας επί του οποίου καταλήξαμε με την ε, Ουκρανία περιγράφεται αναλυτικά στην επιστολή που έστειλαν η Επιτροπή Μάλστρομ και Χόγκεν. Αποτελείται από τρία στοιχεία. Πρώτα απ' όλα οι αυτές οι δύο θεσμολογικές κατηγορίες στις οποίες ε, παρουσιάστηκαν αυτές τις εισαγωγές να ενταχθούν στην ποσόστοση. Δεύτερον, να αυξηθεί η ποσότητα αυτής της ποσότητας, ε, να αυξηθεί η ποσότητα και τρίτον να ε, ξαναεπιβληθούν τα δασμοί MFN ε όταν ξεπερνάται η ποσόστοση. να, να, να εφαρμόζονται λοιπόν δασμοί πλέον ευνοούμενου κράτου όταν ξεπερνάτε ποσόστος. Ε, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο επιλύεται το ζήτημα ικανοποιητικά, ότι είναι εύλογη η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε. Ο κ. μα μας ρώτησε ποια ήταν η εντολή που λάβαμε από το Συμβούλιο. Μπορώ ευχαρίστω, αν θέλετε, να σα δώσω ένα αντίγραφο τη διαπραγματευτική εντολή του Συμβουλίου, αν και αν δεν απατώμε είναι και δημοσίως διαθέσιμο αυτό το έγγραφο. Και μπορείτε εκεί να δείτε τι προβλέπει η εντολή. Η εντολή διαπραγμάτευσης που έλεγε η Επιτροπή από το Συμβούλιο πιστεύω ότι την τηρήσαμε βλαβικά. Τώρα, επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα τρία στοιχεία στη συμφωνία. στο πλαίσιο τη διοργανάτευση αναγνωρίστηκε το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια λογική αναπροσαρμογή τους ποσότητας, της ποσόστοσης ε, και έχω δώσει συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση μου που θα μπορούσαν να σα δώσουν περισσότερε πληροφορίε σε αυτό, εάν θέλετε. Πάντω, η δική μα η ανάλυση έδειξε ότι η ποσόστοση στην οποία είχαμε καταλήξει με την Ουκρανία ήταν μια ποσότητα η οποία θα δημιουργούσε προβλήματα στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν ήταν. Ε, δεν θα δημιουργήσει μάλλον προβλήματα στην ευρωπαϊκή αγορά. Ε, είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει η αγορά μας. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνήσαμε και με τους Ουκρανούς. Τώρα, μια και μιλούμε για εισαγωγέ από την Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, α μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και αντίστροφη κατεύθυνση Δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ουκρανία σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και από πλευρά ποσότητα, ε, το, το, το ισοζύγιο είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ποσότητε που εξάγονται είναι περισσότερε από αυτέ που εισάγονται. Είναι σημαντικό αυτή η συμφωνία να τεθεί σε ισχύ όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Πιστεύω ότι σε αυτό συμφωνούμε οι περισσότεροι. Τώρα δηλαδή που βρέθηκε μια λύση για να κλείσει αυτό το παραθυράκι, είναι προς το συμφέρον όλων μας ε, να την εφαρμόσουμε αυτή τη λύση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Και γι' αυτό το λόγο, σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο επίτροποι σας επέστειλαν αυτή την επιστολή και σας ε, εξηγούν, σας ε, εκθέτουν τα επιχειρήματά τους γιατί χρειάζεται αυτή η εξαιρετική διαδικασία, η έκτακτη διαδικασία να συμφωνήσει δηλαδή το Κοινοβούλιο για ε, μια ε, προσωρινή εφαρμογή. Ο λόγος είναι επειδή προφανώς η ε, το, συνολική συμφωνία, το προσχέδιο της συνολικής συμφωνίας που προετοιμάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα φτάσει αργά έτσι ώστε και άρα δεν θα προλάβει αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή, αυτή τη χρονική περίοδο, την ασαφή, θα αυξηθεί και ο κίνδυνος να υπάρξουν μαζικές εισαγωγές από την Ουκρανία αξιοποιώντας αυτό το παραθυράκι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το κλείσουμε αυτό το παραθυράκι όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Επίσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου. Με αυτά τα επιχειρήματα σας ζητά λοιπόν κατ' η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσετε την έγκρισή σας σε αυτό την ε, τροποποιητική συμφωνία. Κάτι άλλο το οποίο επισήμαναν και πολλοί ευρωβουλευτέ έχει σχέση με τους κανόνες ε, SPS, ε, τους, ε, ασφαλείας. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω ότι οποιοδήποτε εμπορευόμενος από την Ουκρανία που κάνει εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκε και μια συγκεκριμένη εταιρεία, πρέπει να έχει άδεια εξαγωγής προς, προς την Ένωση. Το οποίο σημαίνει ότι οφείλει να τηρεί τους ε, κανόνες, ε, τους υγειονομικούς και φυτογειονομικούς, SPS. Είναι κάτι το οποίο η Γενική Διεύθυνση Σάντε το παρακολουθεί πολύ στενά. Μάλιστα, η Συμφωνία λεφύρων Εμπορίου μα έδωσε τη δυνατότητα να πιέσουμε την Ουκρανία να ευθυγραμμίσει το νομικό τη πλαίσιο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα υγειονομικά και φυτογειονομικά. Έχουν υπάρξει κάποιες ε, συμφωνίες τις οποίες τις παρακολουθούσε η DigiSante και αυτόν τον καιρό προετοιμάζουμε και μια επίσημη συμφωνία η οποία πλέον θα θέτει και ένα χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο η, η Ουκρανία θα πρέπει να εφηγραμμίσει την νομοθεσία της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έχει ήδη πάντως ξεκινήσει να εφηγραμμίζει την νομοθεσία της για τα υγειονομικά η Ουκρανία έχουν ήδη περάσει 200 νόμους ε, στον τομέα αυτό, που είτε και θα έλεγα δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί το έργο που περιμέναμε από τη δικιά του στην πλευρά. Ε, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει αξία το χρονοδιάγραμμα που θα βάλουμε στην ε, μεγάλη, στη Γενική Συμφωνία με την Ουκρανία. Θα το κάνουμε σε κάθε περίπτωση. και θα αξιοποιήσουμε επίση και την εμπειρία και τη βοήθεια ε, από τους συναδέλφου που έχουμε με την ομάδα υποστήριξης της Ουκρανίας, του συναδέλφου, δηλαδή που εκπροσωπούν την Ένωση στο Κίεβο. Ε, στη συμφωνία συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα ε, υγειονομικά, φυτογειονομικά, αλλά επίση και ζητήματα ευζοία των ζώων είναι και αυτό ένα ζήτημα στο οποίο ζητούμε από την Ουκρανία να ευθυγραμμιστεί και να έρθει πιο κοντά στην Ένωση. Αυτά από την πλευρά μου. Τώρα θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου από τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη επίση. Καλησπέρα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σπρίνιερ για να σας δώσει πρόσθετες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω σε δύο ερωτήματα που τέθησαν πρώτο για τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της ποσόστοσης και έπειτα για τους κανόνες προέλευσης του κράτους πληρικών. Οικονομικός αντίκτυπος τώρα. Έχουμε να κάνουμε μια ποσόστοση 50.000 τόνων. Πέρυσι οι εισαγωγές του συγκεκριμένου τεμαχίου είχαν ανέλθει σε 50.000 τόνους περίπου 5.000 τόνοι ανά μήνα. Βλέπουμε ανωδική τάση. Αν υπολογίσετε λοιπόν 5.000 τόνους το μήνα θα δείτε πως το σύνολο θα ανέλθει σε 60.000 τόνους του συγκεκριμένου τεμαχίου. Αν περιορίσουμε δηλαδή την εισαγωγή σε 50.000 τόνους ετησίως θα είμαστε κάτω από το περσινό όριο και σίγουρα κάτω από το προβλεπόμενο όριο για το 2019, για φέτος δηλαδή. Και έτσι λοιπόν θα κλείσει αυτό το παραθυράκι που έμεινε ανοιχτό μέχρι τώρα. Το σύνολο τώρα των εξαγωγών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία είναι 178.000 τόνοι ανά έτος. Πέρυσι δηλαδή ήταν 178.000 τόνοι. Όλες οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών ήταν 123.000 τόνοι. Τι σημαίνει δηλαδή ότι εμείς έχουμε πλεόνασμα εξαγωγών προς την Ουκρανία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες προέλευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες ε, επισήμανσης για την χώρα προέλευσης νοπού και κατεψυγμένου κρέατος πουλερικών. Οι κανόνες αυτοί εγκρίθηκαν το 2013 και ετέθησαν σε ισχύ το 2015. Σύμφωνα με τους κανόνες λοιπόν αυτούς, το νοπό και κατεψυγμένο κρέας πουλερικών που πωλείται πρέπει να αναγράφει την χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής του πουλερικού. Μετά, ο τεμαχισμός σε ύστερο στάδιο που δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην χώρα εκτροφής. Το να βγάλεις ένα κόκαλο από το σφάγιο του ζώου δεν καθιστά το κρέας αυτό ευρωπαϊκής προέλευσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρότι δεν είμαι εμπειρογνώμων για αγροτικά θέματα, δεν με ικανοποιεί η απάντηση. Η νέα ποσόστοση των 50.000 αν δεν κάνω λάθος, η παλιά ποσόστοση ήταν 20.000 τόνοι. Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την αύξηση. Μήπως λόγω του ότι αυτή η μεγάλη κτηνοτροφική εταιρεία μαζί με κάποιες άλλες ε, έκαναν αυτό το κολπάκι με το κόκαλο. Μετά τα πρότυπα. Τα πρότυπα μπορεί να γίνονται σεβαστά ή όχι. Ούτε αυτό είναι σαφές. Ούτε σαφής ήταν και η απάντησή σας. Τώρα, σε περίπτωση καταχρήσεων που θα υπονομεύσουν το σύστημα ε, κατηγοριοποίησης, εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό. Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες έτσι ώστε στην ε, συνάντηση των συντονιστών να αποφασίσουμε για το τι θα κάνουμε. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι έχουμε ενημερωθεί για αυτή την προσωρινή εφαρμογή, αλλά δεν με πείσατε και δεν είμαι σίγουρος ότι θα πείσετε και τους συντονιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, σχετικά με τις ερωτήσεις που κάνατε, πρώτα, ε, το συνολικό ύψος των ποσοστώσεων. Για να είμαι πιο συγκεκριμένος, υπάρχουν δύο ποσοστώσεις 20.000 τόνων στη συμφωνία. Αυτή λοιπόν η πρόσθετη ποσόστοση έρχεται να προσθεθεί σε αυτές τις δύο των 20.000. Όπως είπα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι βασισμένες σε απόρριτα έγγραφα που μας έχουν παραδώσει τελωνιακές αρχές των κρατών μελών. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη μέσω των τελωνιακών του αρχών δεν έχουν πρόβλημα για την κατηγοριοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι ποσοστώσεις είναι νομικά δεσμευτικές για τα προϊόντα αυτά. Δεν μπορούμε λοιπόν να αρνηθούμε ότι υπάρχει ε, νομοδικαίωμα. Έπειτα για τους ε, υγειονομικούς και φυτοϊγειονομικούς κανόνες. Ε, τώρα, το αν τηρούνται. Να σας πω ότι υπάρχει ένα σύστημα μέσω του οποίου χορηγούνται οι άδειες για εισαγωγές από τρίτες χώρες, αλλά οι εισαγωγέ αυτέ πρέπει να συμμορφώνονται πλήρω με του υγειονομικού και φυτοϊγειονομικού κανόνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι συνάδελφοι στη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ έχουν το καθήκον να εντοπίζουν οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας. Δεν έχουμε αναφορές, λοιπόν, για τους κτηνοτρόφους από την Ουκρανία και δεν έχουμε αναφορές ότι έχει υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά την τήρηση των υγειονομικών και φυτογειονομικών κανόνων. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουν οι συνάδελφοι του DG Sante. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Το Φεβρουάριο λοιπόν έγινε ένας έλεγχος από τις υπηρεσίες της Κομισιόν όπου εντοπίστηκαν ιδιαίτερες ε, ε, διαφορές και παραβλέψεις οι οποίες δεν καταγράφηκαν και ε, κατά συνέπεια δεν διορθώθηκαν. Αυτό που λέτε δεν ισχύει λοιπόν. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Θέλετε να ολοκληρώσετε μήπως... Θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Άκουσα τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή και θα το ελέγξω και εγώ, θα ρωτήσω τους συναδέλφους με την ε, Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ. Γίνονται τακτικοί έλεγχοι, όπως αυτός που αναφέρατε. Και οι έλεγχοι αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα διορθωτικά μέτρα για να επιληθούν τα προβλήματα που εντοπίζατε. Ωραία λοιπόν, λέει ο και εγώ αυτό σα συστήνω να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία σα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι. Σα ευχαριστούμε πολύ. Θα συζητήσουμε με τους συντονιστέ το πώ θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Τα σημεία 6β και 7 είναι κυκλισμένων των θυρών. Θα ζητήσω λοιπόν από όσους δεν έχουν το δικαίωμα να παραστούν σε αυτή τη συνεδρία να αποχωρήσουν από την αίθουσα ήσυχα και γρήγορα. Διάλειμμα ενός λεπτού.